Κύριε Προτινόμενο Επίτροπε, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής ε, για αυτή τη μαραθώνια συνεδρίαση. Φυσικά ήταν πολύ έμπειρα με λεξικιωμένα με το θέμα και θα συμφωνείτε ε, κύριε Επιτροπέ ότι αυτή είναι μία από τις πέντε ακροάσεις που συμμετέχουμε αλλά πραγματικά βρίσκεται στο επίκεντρο των αρμοδιοτήτων μας το θέμα της μετανάστευσης του ασύλου, της ε, παράτυπης μετανάστευσης είναι από τα πιο σημαντικά θέματα για μας και γι' αυτό οι συνάδελφοι είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι και ενέκυψα ε, στις λεπτομέρειες του θέματος. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά τα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ και τον προτινόμενο Επίτροπο για την προετοιμασία του για την ακρόαση αυτή. Δεν θα προδικάσω, θα, θα προεξοφλήσω τις περαιτέρω δράσεις, γιατί εναπόκειται στα μέλη της Επιτροπής μέσω των συντονιστών να κρίνουν αυτά που είπατε σήμερα. Και μάλιστα η συνεδρία θα γίνει στις 5 η συνεδρία των συντονιστών για την αξιολόγησή σα. Θα ήθελα εγκατακλείδη να σταθώ σε μερικά πράγματα που είπατε. Αναλάβατε τη δέσμευση να αναθεωρήσετε του μηχανισμού για την λαθρομετανάστευση και τον το σχέδιο της οριζόντιας νομοθεσίας, καθώς θα κάνετε μία ανάλυση της οδηγίας για την κράτηση δεδομένων μετά την πρόσφατη νομολόγια του ΔΕΚ. Επίσης μιλήσετε για μια ενημερωμένη πρόταση για τους φαγγέλους επιβατών, ώστε να γίνονται σεβαστές οι αρχές προστασίας δεδομένων. Επίσης μιλήσετε για τις πρωτοβουλίες της Frontex. Πιστεύω ότι απαντήσατε σήμερα σε σημαντικές προτάσεις και των μελών της Επιτροπής μας, αλλά φυσικά εμείς ε, θα αξιολογήσουμε τη σημερινή ακρόαση με βάση τις ικανότητές σας και με βάση αυτά που μας είπατε σήμερα. Επαναλαμβάνω, η συνεδρία αξιολόγησης θα ξεκινήσει στις 5. Μπορεί να έμειναν κάποιες ε, ερωτήσεις αναπάντητες. Ε, θα ολοκληρώσουμε λοιπόν τώρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και τη συμμετοχή σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στον προτινόμενο επίτροπο για τελικά σχόλια. Τρία λεπτά. Αν επεκταθεί στα πέντε λεπτά θα χάσει όλη την υποστήριξη που κέρδισε νωρίτερα στο κρατήριο. Αν κάνετε κατάχρηση του χρόνου σας θα αποφασίσετε, αλλά ελπίζω να, λάβατε το, να καταλάβατε το υπονοούμενο. Τρία λεπτά είναι αρκετά γιατί είμαστε όλοι εξουθενωμένοι. Τρία λεπτά παρακαλώ για να ολοκληρώσετε και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή αγαπητοί συνάδελφοι Κύριε Προτινόμενο Επίτροπε, σας ακούμε για τα τελικά σχόλια και σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα και καρποφόρα συζήτηση που είχαμε σήμερα. Πραγματικά με διαφωτίσατε σε πολλά θέματα για τα πολύ ευαίσθητα αυτά ζητήματα. Φεύγω από την αίθουσα πιο εμπνευσμένο, πιο ενθαρρυμένο ε, για τα νέα μου καθήκοντα, εφόσον φυσικά ε, επιβεβαιώσετε ως Επίτροπο και αν τελικά επιβεβαιωθεί η υποψηφιότητά μου θα είμαι ο πρώτος Επίτροπος ε, Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τέτοιο θα επικεντρώσω την πολιτική μου πείρα σε τρεις άξονες δράσης. Καταρχήν θα προσπαθήσω να διασφαλίσω, όπως προτείνατε κι εσείς, να εγκρίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ολιστική, σφαιρική και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική που θα στηρίζεται στις αρχές της αναλογικότητας και της αλληλεγγύης, αλλά φυσικά και στην ευθύνη. Επίσης θα αντιμετωπίσω κάποιες σημαντικές προκλήσεις στην ασφάλεια εν των νέων απειλών και των νέων προκλήσεων με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και έχοντα επίγνωση τη ευθύνη ε, τη εξασφάλιση ε, ενό προστατευμένου και ασφαλού περιβάλλοντο για του πολίτε. Επίση, ε, θα συνεχίσω στην πολιτική εσωτερικών υποθέσεων και μετανάστευση σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να έχουμε έναν διαφανή, ειλικρινή και συνεχή διάλογο μεταξύ μας. Θα συνεργαστώ μαζί σας με βάση τη διαφάνεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Thank you. Thank you. Εμείς σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρότινόμενη Επίτροπε. Ακολουθήσατε τη συμβουλή μου. Λήξη της ακρόασης.